υποστηρίξουμε επίσης και τις προσπάθειες της Αμερικανικής κυβέρνησης για να κλείσει επιτέλους ε, η φυλακή του Γκουαντάναμο. Ευχαριστώ Επίτροπε με την δική σας παρέμβαση. Κλείνει η συζήτηση αυτή και θα περάσουμε τώρα στις ψηφοφορίες. Έχουμε 7 προτάσεις ψηφίσματος για το Βιετνάμ. Έχουμε ένα κοινό ψήφισμα από έξι πολιτικές ομάδες. Σχεδόν όλες δηλαδή, πλην της Ανωμένη Αριστεράς. ΕΛΚ, Σοσιαλιστές, άλλοι Πράσινοι, η ΕΦΤ, έχουν το κοινό ψήφισμα. Δεν υπάρχουν τροπολογίες. Ψηφίζουμε λοιπόν το σχέδιο κοινού ψηφίσματος με ονομαστική ψηφοφορία, παρακαλώ. Τύπος είναι φοβερό. Να βάλω και την κάρτα μου, αν με επιτρέπετε. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσαμε όλοι, μάλιστα, πέρας ψηφοφορίας. ομόφωνα εγκρίνεται το κοινό ψήφισμα. Τώρα έχουμε την ψηφοφορία για έξι προτάσεις ψηφίσματος που αφορούν την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Καζαχστάν. Έχουμε μία προφορική τροπολογία. Τροπολογία της κυρίας Ντε Κάιζερ. τεχνικής φύσεως βέβαια, θεωρώ, αλλά η κυρία Ντεκάιζερ θα μας πει. Για να δούμε αν υπάρχει κάποια αντίρρηση, κάποιο πρόβλημα από το σώμα. Παρακαλώ κύριε Ντεκέζερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι στο 1, στην Ανατολική Σκέψη 1, λέγεται σε ό,τι αφορά την επίσκεψη της κυρίας Άστον στην Κεντρική Ασία και το Καζακστάν ότι δεν έκανε καμία δήλωση μετά. Λέει, λαμβάνοντα υπόψη ότι δεν εξέδωσε καμία δήλωση για το θέμα αυτό, στο N ή Ι Δέλτα ελληνικό. Εγώ θα έλεγα να προσθέσουμε μετά για το, από το, για το θέμα αυτό στη διάρκεια της επίσκεψης αλλά μετά, το Δεκέμβριο 2012. Δηλαδή εννοούμε ότι ναι, δεν έκανε δήλωση το Νοέμβριο στη διάρκεια τη επίσκεψη, έκανε όμω δήλωση το Δεκέμβριο του 2012. Ευχαριστώ, Βερονίκη Πρόεδρο. Δεν βλέπω να υπάρχει κάποια αντίρρηση, άρα μπορούμε να ψηφίσουμε το κείμενο του κοινού ψηφίσματος με την προσθήκη αυτή. Νομίζω ναι ότι ψηφίζουμε ονομαστικά και σε αυτή την περίπτωση. Ωραία, άρχεται η ψηφοφορία λοιπόν. Ψηφίσαμε όλοι. Τώρα ναι. Ψηφίσαμε όλοι. Πέρασε ψηφοφορίας. Βλέπετε το αποτέλεσμα στην οθόνη. Εγκρίνεται το κείμενο με πάρα πολύ μεγάλη πλειοψηφία. Τα πρακτικά θα τεθούν υπόψη του Κοινοβουλίου για έγκριση στην επόμενη ε, σύνοδο. Τα ψήφισματα που επεγκρίθηκαν θα ε, διαβιβαστούν στα άτομα και τα ε, όργανα τη φορή που αναφέρονται σε αυτά τα ψηφίσματα. Πριν ολοκληρώσουμε, σα επαναλαμβάνω αυτό που είπα και πριν, ότι ο κύριο Πόσε